εδώ η συζήτηση αυτή. Τα πρακτικά, τα συνοπτικά θα διανεμηθούν στην αρχή της επόμενης συνόδου ε, και αν δεν διαφωνεί κανείς τα ε, εγκεκριμένα πρακτικά θα διαβιβαστούν και αποφάσεις του Κοινοβουλίου θα διαβιβαστούν αρμόδιως. Διακόπτεται η σύνοδος. Και σας εύχομαι καλή επάνωδο και με ασφάλεια στις χώρες σας. Ευχαριστώ πολύ.